Καλησπέρα κύριε και κύριοι, συνάδελφοι. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για την ανάπτυξη της πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών βάσει του άρθρου 11 παραγράφου 4 της Συνθήκης της Ένωσης. Δώστε μου την άδεια σας παρακαλώ να καλωσορίσω με μεγάλη αγάπη μια ομάδα από την περιφέρειά μου, την Λαμάντσα, Καστίγια Λαμάντσα, που επισκέπτονται αυτές τις ημέρες τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Καλώς ήρθατε. Για το ξεκίνημα της συζήτησης αυτής δίνουμε το λόγο στον Υπουργό κ. Λόπεθ Καρύγου εξ του Συμβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο που ξεκίνησε την πρωτοβουλία να προχωρήσει στην συζήτηση αυτή για ένα από τα πιο σημαντικά πιστεύω θέματα της συνθήκης από την οπτική γωνία της δημοκρατίας και της ανάπτυξης της Ένωσης και της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού ιδεόδους μεταξύ των πολιτών που μπορούμε να δούμε σε ένα τόσο σημαντικό κείμενο που ανοίγει μια νέα φάση στην Ένωση. Όπως γνωρίζετε, μιλώ για το θέμα της πρωτοβουλία πολιτών. Τη δυνατότητα δηλαδή ένα εκατομμύριο πολιτών τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διάφορες χώρες της Ένωσης, να υπογράψουν μια νομοθετική πρωτοβουλία που λογικά απευθύνεται προς την Επιτροπή, τίθεται προς την Επιτροπή που είναι το κοινοτικό όργανο που έχει την ικανότητα νομοθετικής πρωτοβουλίας, την αρμοδιότητα νομοθετικής πρωτοβουλίας. Η πρωτοβουλία των πολιτών αποτελεί μια σαφή, πολύ σαφή προτεραιότητα της Προεδρίας Συμβουλίου. Πολύ σαφή. Και τούτο διότι θεωρούμε ότι αποτελεί προτεραιότητα και της Ευρώπης. Όταν μια χώρα προεδρεύει του Συμβουλίου της Ένωσης, Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να αναπτύξει τους δικούς της στόχους, ε, να προωθήσει τους δικούς της στόχους, ως χώρα απλά. Πρέπει να μπορεί ταυτόχρονα και να εκπροσωπεί τους στόχους της Ευρώπης. Η πρωτοβουλία πολιτών δίνει στους πολίτες της Ένωσης ένα σημαντικό δικαίωμα και αποτελεί αυτό ένα μεγάλο στόχο της Ένωσης και αυτό είναι προτεραιότητα και της Ισπανίας και της Ισπανικής Προεδρίας και της Ευρώπης πρέπει να είναι. Οι πολίτες περιμένουν να προχωρήσει η συνθήκη της Λισαβόνας στο συντομότερο δυνατό μετά από 8 χρόνια χαμένου χρόνου σε θεσμικές αβεβαιότητες. Πρέπει να κερδίσουμε τον χρόνο αυτό και να απαντήσουμε κυρίως στους πολίτες. Αυτό που θέλουν είναι η συμμετοχή. Δηλαδή το να υπάρξει μια νέα ισορροπία μεταξύ της Ευρώπης που οικοδομείται κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα από πάνω προς τα κάτω, έστω και αν είναι δημοκρατική, προς μια Ευρώπη που χτίζεται από κάτω προς τα πάνω. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Γιατί αποτελεί απόδειξη θα αποτελεί απόδειξη μάλλον της πολιτικής βούλησης των κυβερνήσεων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δοθεί στους πολίτες φωνή και ικανότητα συμμετοχής και για να σταματήσουμε κάτι που δυστυχώς συμβαίνει στην Ένωση ο πολιτικός διάλογος να είναι κατά βάση ένας εθνικός, ενδογαμικός διάλογος. Στις Βρυξέλλες, εδώ, κάνουμε ευρωπαϊκό διάλογο. Σε όλες τις χώρες της Ένωσης κυριαρχεί η εθνική συζήτηση. Η συζήτηση για εθνικά ζητήματα, όχι για την Ευρώπη. Και η πρωτοβουλία πολιτών είναι ένα εξαιρετικό μηχανισμός για να απεγκλωβίσουμε στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών την δυνατότητα αυτή και να την μετατρέψουμε, να μετατρέψουμε το διάλογο σε έναν πραγματικά ευρωπαϊκό διάλογο να εμφανίσουμε έναν ευρωπαϊκό διάλογο σε όλες τις χώρες, όχι μόνο έναν εθνικό. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, θεωρήσαμε την πρωτοβουλία πολιτών ως μία πρωτοβουλία, μία προτεραιότητα, συγγνώμη. Θεωρούμε ότι από τη στιγμή που η Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο κανονισμού, και ευχαριστούμε τον Επιτροπή, διότι ιδιαίτερα τον, κύριο, τον πρώτο, τον κύριο Μπαρόζο και τον αντιπρόεδρο κύριο Σέρκοβιτς. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί έδειξαν ότι αποτελεί το θέμα αυτό προτεραιότητα και της Επιτροπής στο πρόγραμμα εργασία της Επιτροπής. Την ευχαριστούμε λοιπόν, τους ευχαριστούμε διότι έχουμε ένα κείμενο που θα μπορέσει να έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή πριν ολοκληρωθεί η, το εξάμεινό μας. Προφανώς θα πρέπει να δούμε τις διάφορες πτυχές που πρέπει να λυθούν, θέματα τεχνικά, θέματα πολιτικά, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβεί κάτι τέτοιο. Εμείς λοιπόν από την άτυπη συνάντηση υπουργών ευρωπαϊκών υποθέσεων στην Λαγκράνχα, θα το, το, το, το, θα το θυμίσει ο κύριος ε, και με την κυρία Μάλσο γιατί δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η νέα επιτροπή και στη συνάντηση που είχαμε στη Μαδρίτη με την ε, έναρξη, με την ε, ανάληψη των καθηκόντων της νέας επιτροπής έχουμε δείξει ότι μας ενδιαφέρει να προχωρήσουμε την πρωτοβουλία αυτή και ζητώ από εσά κυρίες και κύριοι βουλευτές να δείξετε το μέγιστο δυνατό ενδιαφέρον προς την πρωτοβουλία αυτή. Ξέρω ότι το κάνετε, αλλά θέλετε, θα ήθελα να ε, προχωρήσετε γρήγορα κάτι που την χάνει της γενικής συνένεσης. Λόγω των συζητήσεων που είχαμε, που έχουμε στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ειδικότερα, για να προχωρήσει στην υλοποίηση ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία για τους Ευρωπαίους πολίτες στη νέα αυτή φάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Υπουργό για την Επιτροπή. Το λόγο έχει τώρα ο Αντιπρόεδρος και φίλος κύριος Σεύκοβιτς. Ευχαριστώ, να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έθεσε στην ημερήσια διάταξη το πολύ σημαντικό αυτό σημείο. Να ευχαριστήσω προσωπικά τον αγαπητό φίλο Διέγκο και την Ισπανική Προεδρία που τοποθέτησαν το θέμα αυτό και στην ε, κορυφή των προτεραιοτήτων της Ισπανικής Προεδρίας. Γιατί νομίζω ότι το, αυτό θα αλλάξει το πώς ασκείται η πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ως τώρα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα βασιζόταν στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Και αυτό αντικατοπτριζόταν και στην συνθήκη της Λισαβόνας, όπου ήταν σαφές ότι ενισχύονται οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες των ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι θα συμμετέχουν πιο έντονα και τα εθνικά κοινοβούλια. Άρα χρειαζόταν και η πιο έντονη συμμετοχή των πολιτών και με το εργαλείο αυτό της συμμετοχικής δημοκρατίας. Έγινε μια συζήτηση ότι το ένα δεν αποκλείει το άλλο και πραγματικά το πιστεύω αυτό γιατί θεωρώ ότι και τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν ε, εκφάνσεις της συμμετοχικής δημοκρατίας και βοηθάει το ένα το άλλο για τη δημιουργία πραγματικά ευρωπαϊκού πολιτικού σκηνικού. Θεωρώ ότι αυτό υπογραμμίζει ακόμα πιο πολύ τη σημασία του Ευρωπαίου πολίτη. Όπως είπε και ο Ντιέγκο ήδη, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια πιο ισχυρή, καλύτερη συζήτηση πανευρωπαϊκή, πιο πολύ για ευρωπαϊκά θέματα, όχι μόνο για εθνικά θέματα, το οποίο βλέπουμε ότι συμβαίνει σήμερα στις πρωτεύουσε των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν και είναι ευγνώμων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, δουλειά που έχει κάνει σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία των πολιτών. Και το ψήφισμα της 7ης Μαΐου του περσινού έτους ήταν πάρα πολύ σημαντικό ως πολιτική καθοδήγηση για την προετοιμασία της πρωτοβουλίας αυτής. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν προετοιμάζει τέτοια σημαντικά ε, νομοθετήματα θέλει πάντα να έχει και τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στο βαθμό του δυνατού. Γι' αυτό λοιπόν και διοργανώθηκαν δημόσιες συζητήσεις βάσει της Πράσινης Βίβλου που εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 2009. Θα πρέπει να διευκρινίσω ότι μας προκάλεσε θετική έκπληξη οι απαντήσεις ε, που λάβαμε. Λάβαμε, πιο, λάβαμε περισσότερες από 300 απαντήσεις από διάφορους ε, πολίτες, τοπικές αρχές, ε, οργανώσεις, από εθνικά κοινοβούλια. Αξιολογήσαμε τις απαντήσεις που λάβαμε. Συμπληρώσαμε και ολοκληρώσαμε τη διαδικασία δημοσίων διαβουλεύσεων με μια δημόσια συζήτηση στις Βρυξέλλες στην οποία συμμετείχαν 150 και πλέον ε, αρμόδιοι φορείς και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συνοψίσω λοιπόν τη συζήτηση αυτή. Θα πρέπει να πω ότι πολλά καινοτομικά στοιχεία παρουσιάστηκαν, πολλές πρωτότυπες ε, προτάσεις υποβλήθηκαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα βασικά συμπεράσματα ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την εφαρμογή Τη πρωτοβουλία αυτή το συντομότερο δυνατόν, ότι θα θέλα να είναι όσο πιο φιλική αν θέλετε προς το χρήστη γίνεται αυτή η διαδικασία, κατανοητή, προσβάσιμη και απλή. Θα συμφωνήσετε φαντάζομαι ότι πρόκειται για σαφείς ε, και ξεκάθαρες παράμετρους οι οποίες θα πρέπει να ορίσουν την ε, κατάρτιση της νομοθεσίας γιατί μόνο έτσι θα χρησιμοποιήσουν οι πολίτες ε, το εργαλείο αυτό για καλύτερη και πιο στενή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με του Ευρωπαϊκού θεσμού. Μετά λοιπόν τα αποτελέσματα και τα πορίσματα των διαβουλεύσεων, κοιτώντα και τι προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει στην παρούσα φάση την πρόταση την οποία θα υποβάλει. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να την υποβάλουμε μέχρι Μαρτίου. Να σας πω επίσης ότι αυτό δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς ε, την ε, έντονη ενθάρρυνση της Ισπανικής Προεδρίας, γιατί είναι σαφές ότι θα πρέπει να σεβαστούμε το γεγονός ότι αυτό αποτελεί προτεραιότητα της Ισπανικής Προεδρίας. Ξέρω άλλωστε πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό για την Ισπανική Προεδρία. Θέλει να το ολοκληρώσει πριν το τέλος ε, της Προεδρίας της. Να ευχαριστήσω λοιπόν και θεωρώ ότι χάρη στην ηγεσία του Κοινοβουλίου και της ε, Ισπανική Προεδρία θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την, ε, το μέσο αυτό πριν από την πρώτη επέτειο τη θέση ισχύ τη συνθήκης της Λισαβόνας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και σε και τώρα για να δούμε του ε, αγορητέ των κοινοβουλευτικών ομάδων. Πρώτα-πρώτα για δύο λεπτά έχει το λόγο ο κύριο Ίνιγο Μέντε Τεβίγκο για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε εδώ. Σε αυτό το ίδιο ημικύκλιο πριν από 7 χρόνια όταν είχε ολοκληρωθεί η συντακτική, συνταγματική διαδικασία και συνέλευση σε συνεργασία με τους βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων Λαμασούρ και Γιούργεν Μάιερ είχαν υποβάλει και την πρόταση για αυτή την ε, πρωτοβουλία που τελικά κατέληξε στην συνθήκη που, που ισχύει στην νίκη τη Λισαβόνα και όπω είπε ο Σεύκοβιτ, αυτό είναι συμμετοχή η δημοκρατία, συμμετοχή των Ευρωπαίων. Ε, άρα θα πρέπει η συμμετοχή μα οδηγεί στο να είμαστε περισσότερο Ευρωπαίοι και να ανάγονται τα θέματα και συζητήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μα είπε όμω ε, ο κύριο Επίτροπο ακριβώ τι λεπτομέρειέ του πώ θα, θα, θα, θα ε, υλοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία φτάσαμε μέχρι την πηγή δεν ήπιαμε νερό γιατί θα πρέπει να δούμε πώς μετά από αυτές τις εξαγγελίες πώς θα μπορέσει ακριβώς χωρίς κανείς να έχει πτυχία πνευματικά θα μπορέσει να συμμετάσχει πώς δηλαδή θα γίνει αυτή η συνεργασία των ευρωπαϊκών οργάνων και των ε, εθνικών αρχών γιατί κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό ρόλος των εθνικών αρχών. Κατά τρίτο λόγο, αυτό το οποίο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσαμε να διαπαιδαγωγήσουμε τον κόσμο για να του εξηγήσουμε πώ μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία, ούτω ώστε να μην πέσει στο κενό και απογοητευτούμε. Ε, είχαμε την πρωτοβουλία Intermedia, συλλογή υπογραφών, ούτω ώστε να είναι δυνατόν να σταματήσουμε μετακινούμεθα ω κοινοβούλιο και να έχουμε μόνο μία έδρα, όμω είπαμε ότι αυτό δεν γίνεται, χρειάζεται αναφιέρωση των συνθήκων. Δεν γίνεται τον αυτό να γίνει με δημοψήφισμα και με τέτοιου είδου λαϊκέ πρωτοβουλίε. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να διαπαιδαγωγήσουμε τον κόσμο. Είναι μια πρωτοβουλία που ε, το ΕΛΚ το ενθουσιάζει και θεωρούμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να ε, τονώσουμε το συνέστημα του ανήκειν στους Ευρωπαίους ως προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για δύο Ο κύριος για τον των Σοσιαλιστών ευχαριστώ. Πρόεδρε, πάρα πολύ χαρά μας δημιουργεί αυτό το οποίο είπε ο κ. Σεύκοβιτς ε, και ο οποίος καλωσόρισε γιατί μας είπε ότι στις 31 Μαρτίου ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εγκρίνει αυτό το σχέδιο κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό, να γίνει και συγχαρητήρια στην Προεδρία και στην Κομισιόν και στον κύριο Επίτροπο συγκεκριμένα για την προώθηση αυτής της πρωτοβουλίας και μια που κατάφεραν να συμφωνήσουν τα δύο θεσμικά όργανα και να κατεβάσουν ενώπιον μας αυτή την πρόταση που είναι σημαντική γιατί νομίζω ότι έτσι θα αναβαθμιστεί η δημοκρατική νομιμότητα του Κοινοβουλίου γιατί κατά αυτόν τον τρόπο ο Ευρωπαίος μπορεί να έχει προσβασιμότητα άμεση στο Κοινοβουλίο και όχι μέσω των κομμάτων. Ο ίδιος ο πολιτή μπορεί να έρθει εδώ και αυτό το καταφέραμε με, με, με ένα απλό νομοθέτημα, ούτω ώστε να μπορεί να έχει περισσότερη δημοκρατική νομιμότητα το Κοινοβούλιο, γιατί η βάση του Ευρωπαϊκού Οράματο είναι ο πολίτης, είναι ο Ευρωπαίος, είναι ο βασικός άξονας του Ευρωπαϊκού Οράματο και άρα αυτός πρέπει να πρωταγωνιστεί. Επίσης, νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε καλύτερη λειτουργία καλύτερη σχέση ε, θεσμικών οργάνων και των Ευρωπαίων, κατά το οποίο πάντοτε το λέμε αλλά δεν γίνεται. Ε, υπάρχει προσέγγιση, υπάρχει κατανόηση του τι ωφελεί να υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι χρησιμεύει. Τώρα, θα, συμβούσουμε με τον κύριο Μέντες Δεδίκο σε κάποιες προτάσεις που θέλω να κάνω για να βοηθήσω Νομίζω ότι θα πρέπει να προβλέπεται ένα κείμενο, ένα νόμο που να είναι ευέλικτο, τόσο ώστε να επιτρέπει την άσκηση αυτού του δικαιώματο. σε όσο γίνεται περισσότερου. Γιατί άμα κάτσουμε να λέμε σε ποιε χώρε τι θα γίνει, ε, η κάθε χώρα πόσε υπογραφέ θέλει. Ε, θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι να διευκολύνουμε την ε, υλοποίηση αυτή τη πρωτοβουλία και θα πρέπει αυτό να είναι ξεκάθαρο. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε απογοήτευση στι προσδοκίε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προλυάνει το έδαφος και να δει τι γίνεται αν κάποια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να ευδοκιμήσει εάν είναι βάσιμο και αυτό πριν γίνει η συλλογή των ε, υπογραφών ούτως να μην απογοητεύσουμε κανένα άρα να είμαστε σαφείς και ευέλικτοι για αυτή την υπόθεση Βεβαίω και σα χαίρω ακόμη μια φορά. Ευχαριστούμε κύριε Χάρη. Και τώρα για του ελευθέρου έχει το λόγο η κυρία Χατενμάκη. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η πρωτοβουλία των πολιτών είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση που πρόθεσε η συνθήκη της Λισαβόνας. Ενισχύει την απευθείας επιρροή των πολιτών στα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα. Προφανώς είναι ένα μικρό βήμα και δεν είναι εύκολο να, μαζέψει κανείς ένα εκατομμύριο υπογραφές. Όταν όμως το πετύχει, αυτό που κάνει κάποιος είναι απλά να μπορέσει να ζητήσει από την Επιτροπή να αναλάβει δράση και η Επιτροπή εν τη σοφία της αποφασίζει κατά πόσον ή όχι θα δώσει συνέχεια στην πρόταση. Για να πετύχει η πρωτοβουλία των πολιτών μπορεί ενδεχόμενα να προχωρήσουμε σημαντικά στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Τώρα που ετοιμάζουμε το νομοθετικό πλαίσιο για την πρωτοβουλία των πολιτών πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η διαδικασία θα είναι ξεκάθαρη, οι κανόνες σαφή και κατανοητοί για τους πολίτες. Δεν θέλουμε προς Θεού να δημιουργηθούν ψευ, ψευδείς ελπίδες ή να υπάρξουν παρανοήσεις. Πιστεύω ότι η διαδικασία εξέτασης εξ άντε αξίζει να μελετηθεί διότι μπορεί να έχει θετικές συνέπειες. Δεν είμαι όμως βέβαιη κατά πόσον μπορεί να υπάρξει, είναι σκόπιμο να υπάρξει μια αρνητική απάντηση σε πολύ πρώιμο, πρώιμο σε πολύ πρώιμη χρονική στιγμή. Επίσης, πιστεύω ότι το όριο θα πρέπει να είναι το 1 τέταρτο των κρατών μελών για την πρωτοβουλία. Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να θέτει εμπόδια στην πρωτοβουλία των πολιτών. Πρέπει να υπάρχει ένα κείμενο σαφές και απλό και ελπίζω να υπάρξουν πολλές τέτοιε πρωτοβουλίες και να τις δεχθεί η Επιτροπή. Για τους πράσινους και για τρία λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Χέφνερ. Σας ευχαριστώ αξιότιμη πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Διέγκο, ε, κυρία Επίτροπε, έχουμε μια τεράστια ευκαιρία αυτή τη στιγμή, μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη. Για την κοινή αυτή η Ευρώπη που ξεκίνησε με συνθήκες μεταξύ κρατών, δηλαδή με ένα κλασικό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, όπου ουσιαστικά ο πολίτης ήταν θεατής. Τώρα να κινηθούμε προς μια Ευρώπη των πολιτών. Αυτό που συζητάμε εδώ σήμερα είναι το πρώτο εργαλείο μιας άμεσης συμμετοχής των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σαφές τι σημαίνει αυτό, τι ευκαιρίες συνεπάγεται, κυρίως για τη δημιουργία σταδιακά μιας ευρωπαϊκής κοινή γνώμης, ε, την οποία χρειάζεται η Ευρώπη αυτή, γιατί ακόμα στην ε, Γαλλία, στην Πορτογαλία, στη Γερμανία συζητιόνται λίγο πολύ ξεχωριστά εθνικά θέματα. Σε ό,τι αφορά τους πολίτες δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή ε, συζήτηση, ευρωπαϊκός διάλογος, αλλά αυτό θα μπορούσε να προεθωθεί με την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών προκειμένου να ξεπεραστεί η αίσθηση του πολίτη ότι απέχει τόσο πολύ πια ε, απέχουν τόσο πολύ οι από τον ίδιο. Δημιουργούμε ένα πρώτο εργαλείο που δίνει ένα τρόπο συμμετοχής των πολίτη, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα διαμορφώσουμε το εργαλείο αυτό. Το κατά πόσο θα υπάρξει επιτυχία δεν έχει ακόμα αποφασιστεί αυτό, εξαρτάται από τη διαμόρφωση του εργαλείου αυτού. Και καταλαβαίνω φυσικά ότι δεν μπορείτε σήμερα να μας ε, παρουσιάσετε τις λεπτομέρειες του εργαλείου αυτού, γιατί δεν έχουν αποφασιστεί ακόμα, αλλά έχουμε κάποια κοινά στοιχεία τα οποία θέλουμε, κάποια στοιχεία που μας απασχολούν όλους. Να τονίσω το εξή, Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ή τουλάχιστον αυτό που θα αποφασίσουμε ως νομοθετική πρόταση στο τέλος δεν θα πρέπει να περιέχει μόνο εμπόδια τα οποία θα πρέπει ε, να τηρούν οι πολίτες. Θα πρέπει να περιέχει και να προβλέπει πώς θα επεξεργάζεται με σοβαρό τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια τέτοια πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί είναι πάρα πολύ απογοητευτικό αν μια τέτοια πρόταση έχει καταφέρει να μαζέψει ένα εκατομμύριο υπογραφές δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να το ξεχνάμε. Χρειαζόμαστε τρία επίπεδα τυπικών προδιαγραφών. Πρώτον θα πρέπει να συλλεχθούν οι υπογραφές. Κατά δεύτερον είναι, θα πρέπει να έγκυται στον τομέα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τέλος, θα πρέπει να γίνεται και ένας έλεγχος επί του περιεχομένου. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να εμπλακεί πιο πολύ και να συμμετάσχει ο πολίτης, να τους καλέσουμε και να μην τους παρουσιάζουμε ε, de facto αποτελέσματα. Και μία δεύτερη παρατήρηση, επιτρέψτε μου, ένα τρίτο, το 1 τρίτο, το εννέα κράτη-μέλη τα οποία θα πρέπει να εκπροσωπούνται, μου φαίνεται ότι είναι υπερβολικά υψηλό ποσοστό. Εμείς ήμασταν υπέρ του ενός τετάρτου των κρατών μελών και στις ε, συζητήσεις είχα προτείνει να λάβουμε ε, υπόψη και το μέγεθος του κράτους μέλους, γιατί έχει διαφορά αν μιλάμε για μεγάλος ή μικρό κράτος μέλος. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ για τα υπόλοιπα σημεία, δυστυχώς λόγω χρονικών περιορισμών, αλλά θα ήθελα διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ξεπεράσετε την ώρα σας. Για τους μεταρρυθμιστές και συντηρητικούς, ο κύριος Καμάλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Πολύ καλωσορίζουμε όποια πρωτοβουλία μειώνει τις εξουσίες από την Ένωση και τις περνάει στον πολίτη ξανά. Θα ζητήσω λοιπόν σε μία διάσταση μεγαλύτερη ευελιξία. Γιατί να αποφασίζουμε εμείς τους λόγους για τους οποίους μπορεί να ξεκινήσει ο πολίτης μία πρωτοβουλία. Ας την ξεκινήσει και ας παρουσιάσουμε ο πολίτης και ας παρουσιάσουμε τις απόψεις μας όταν παρουσιαστούν. Εμείς δεν θα πρέπει να προδικάζουμε αλλά να απαντάμε. Ας αντιμετωπίσουμε τους πολίτες ευθεία, ευθέως. Ένα θέμα θέλω να θέσω. Την διαφάνεια. Δύσκολα οι πολίτες μόνοι τους θα μπορούν να καλύψουν τις υπογραφές αυτές. Θα έπρεπε λοιπόν οι οργανώσεις που συγκεντρώνουν τις υπογραφές να είναι διάφανες για τους λόγους και τη χρηματοδότησή τους. Να μην ζητούν ε, να είναι πραγματικές πρωτοβουλίες των πολιτών και όχι πρωτοβουλίες οργανώσεων ή της κοινωνίας των πολιτών και των νοικίων. Ευχαριστώ. Για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά το λόγο έχει ο κ. Σάντερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έλλειψη εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ένωση είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε. Η μικρή συμμετοχή στις ευρωεκλογέ δείχνει ξεκάθαρα την έλλειψη εμπιστοσύνη των πολιτών. Αν την πρωτοβουλία των πολιτών την ερμηνεύσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε λίγοι να τη χρησιμοποιήσουν, θα επιδεινώσουμε την κατάσταση. Δεν θα πρέπει οι κανόνες για την πρωτοβουλία των πολιτών να είναι εξαιρετικά αυστηροί. Πρέπει να είναι προφανώς ένα σημαντικό ευρωπαϊκό θέμα, αλλά μπορεί να υπάρξει ένα εκατομμύριο υπογραφέ από μικρό αριθμό κρατών μελών. Ω μέλη του Κοινοβουλίου θα πρέπει να φροντίσουμε το ώστε η πρωτοβουλία των πολιτών να αντιμετωπίζεται με σοβαρό τρόπο και να ε, εξασφαλίσουμε ταυτόχρονα ότι μπορεί να, θα μπορεί να προχωρήσει και για το θέμα αυτό μπορεί να γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια αλλά μια συζήτηση που θα δείξει που θα δίνει μια κατεύθυνση και για το επίμαχο ζήτημα δείχνοντας έτσι ότι πραγματικά τιμούμε την έννοια της πρωτοβουλίας των πολιτών. Για την ολοκλήρωση της σχετικής συζήτησης ο κύριος Βανέκε για ένα λεπτό εξ ονόματος των μη εγγεγραμμένων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ω τώρα άκουσα με μεγάλη δυσπιστία τα όσα υπόθηκαν. Ξέρουμε από την εμπειρία των δημοσκοπήσεων στη Γαλλία και στην Ολλανδία και από το τελευταίο στην Ιρλανδία. Ξέρουμε ποια είναι η γραφειοκρατία και η αντίδραση του κόσμου στη γραφειοκρατία. Τι προβλέπει αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών ουσιαστικά αποτελεί, αν θέλετε, ένα παραπέτασμα που θα έπρεπε να παραπλανήσει τον Ευρωπαίο πολίτη στη συνθήκη της Λισαβόνας χωρίς ουσιαστικά να δίνει μεγαλύτερη συμμετοχή στην διαδικασία αυτή της λήψης αποφάσεων. Ουσιαστικά ε, περιλαμβάνονται εμπόδια, γραφειοκρατικές ε, γραφειοκρατικά εμπόδια και στην περίπτωση που τελικά υπερπληκτούν όλα αυτά θα είναι το ίδιο το αποτέλεσμα. Αυτό που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη είναι δεσμευτικά ε, δεσμευτικές δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την προσχώρηση της Τουρκίας. Εκεί θα ήταν χρήσιμη η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών και δυστυχώς αποτελεί αυτό μια καρικατούρα και μόνο. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε έτσι τον κύκλο των αγωγητών για τις πολιτικές ομάδες και ξεκινούμε με τους αγωγητές ε, με τους, ε, σε ατομικό επίπεδο. Για δύο λεπτά ο κύριος Καζίνη, πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Δέχομαι θετικά τις δηλώσεις ε, του Υπουργού κ. Γκαρίγκο και του Επιτρόπου Σεύκοβιτς ε, που για πρώτη φορά με τη συνθήκη της Λισαβόνας καθιερώνει την πρωτοβουλία των πολιτών που μαρτυρεί την ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού λαού. Ένα, άλλωστε, μία από τις βασικές επικρίσεις κατά της Ένωσης είναι ότι δεν είναι μια πραγματικά δημοκρατική δομή. Η συνθήκη της Λισαβόνας προσπάθησε να μειώσει το δημοκρατικό έλλειμμα με πολλούς τρόπους, μεταξύ αυτών και η πρόβλεψη της δυνατότητας ένα τουλάχιστον εκατομμύριο πολιτών να μπορούν να υποβάλουν μια νομοθετική πρωτοβουλία το νέο θεσμικό πλαίσιο ωστόσο γεννή σοβαρό πρέπει να έχει κάποιες ε, νομικές ε, ρυθμίσεις. Δεν πρέπει να ταυτίστε με μια αναφορά από άτομα. Θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορά μεταξύ τους. Θα πρέπει κατά συνέπεια να έχει συγκεκριμένη ρύθμιση, συγκεκριμένους κανόνες που θα ε, αποτρέπουν τις καταχρήσεις αλλά θα επιτρέπουν ταυτόχρονα έναν ουσιαστικό και επαληθεύσιμο ε, τρόπο λειτουργία τη διαδικασία αυτή. Η πρωτοβουλία αυτή, ωστόσο, που στο άρθρο 11 τη συνθήκη τη Λισαβόνα, περιέχει και ένα συμβολισμό. Το δημοκρατικό έλλειμμα καταπολεμάται όχι με την, ε, μόνο με την αποφασιστική ε, αρμοδιότητα των εκπροσώπων του λαού, αλλά από την ύπαρξη καταρχήν ενός ευρωπαϊκού λαού που δεν το άθροισμα των εθνικών λαών. Γι' αυτό θεωρούμε πολύ σημαντικό στο πλαίσιο αυτό δύο πράγματα. Πρώτον, το θέμα. Όπως το είπε κάποιος, το θέμα πρέπει να είναι ευρωπαϊκό. Δεύτερον, η κατανομή του ελάχιστου αριθμού υπογραφών σε έναν σημαντικό αριθμό κρατών μελών με ένα αντίστοιχο κατάλληλο προτυπώ σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας. Εύχομαι το νέο νομοθετικό πλαίσιο να επιτρέψει σε Ισπανούς, Γάλλους, Γερμανούς, Ιταλούς, αλλά κυρίως σε Ευρωπαίους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ευχαριστώ κύριε Καζίνη. Η κυρία Γκουρμάη, για ένα λεπτό. Η πρωτοβουλία για τον Ευρωπαίο πολίτη είναι μια καινοτομία βασική, πολύ σημαντική συνθήκη της Λισαβόνας. Γιατί έτσι αναβαθμίζεται η άμεση δημοκρατία στην Ευρώπη θα πρέπει να καταληφθούμε αυτέ τι δυνατότητε όσο γίνεται περισσότερο και θα πρέπει έτσι να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία του θεσμού. Και γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν τα εξή δύο. Βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να αλλά τα βασικά είναι πρώτα-πρώτα ότι οι υπογραφέ θα πρέπει να είναι δυνατόν να διασταυρωθούν και να επαληθευτούν και να μην έχουμε κάποια προβλήματα από την πολυνομία που υπάρχει γιατί κάθε χώρα έχει τα δικά της. Δηλαδή άρα να έχουμε κάποιο είδου κοινή νομική πλατφόρμα. Δεύτερον, το παραδεκτό, το βάσιμο, θα πρέπει να υπάρχει εξέταση για να κρίνεται η συνέχεια. Θα πρέπει να δούμε ποιες αρχές θα υιοθετηθούν και θα πρετανεύσουν, να μην έχουμε αντιφάσεις και πρωτοβουλίες που μία να ακυρώνει την άλλη. Άρα θα πρέπει το νωρίτερο δυνατόν να ε, ρυθμίζουν λεπτομέρειε, τόσο ώστε να εφαρμοστεί πλήρω αυτή η ιδέα και να δούμε μετά τη συνάντηση που θα κάνετε τι θα κάνει η Κομισιόν, τι μέτρα θα πάρει όσον αφορά αυτά που είπαμε, δηλαδή την εξακρίβωση των υπογραφών και την κρίση του παραδεκτού και βάσιμου. Επομένω θα προχωρήσουμε σε ένα κείμενο και δικό μα εδώ έκθεση ε, για την καλύτερη προσέγγιση και νομίζω ότι για εμεί εδώ πέρα τον Ευρωπαίο πολίτη εκπροσωπούμε. Άρα θα πρέπει να δούμε πώ θα μπορέσουμε το μήνυμα που θα στείλουμε να είναι όσο γίνεται πιο αποφασιστικό. Νομίζω ότι πάρα πολύ καλά τα πάει η, Ισπανική Προεδρία όπω και η υπόλοιπη Τρόικα, η Βελική και η Ουγγρική Προεδρίας. Καλά τα πάτε, συνεχίστε. Ένα μισή λεπτό, λέει ο Πρόεδρος για την κυρία Γουόλης την Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο έχει τεράστιο δυναμικό και θα μπορούσε να αποστείλει ένα πολύ σημαντικό και χειρό δημοκρατικό μήνυμα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στη χώρα μου, αν θέλει κάποιος να ε, προωθήσει νομοθετική πρωτοβουλία, θα πρέπει να βρει ένα βουλευτή, θα πρέπει αυτός ε, να σταθεί πάρα πολύ τυχερός και να τον εγκρίνει το αίτημά του και η κυβέρνηση η εκάστοτε. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το εργαλείο το οποίο ετοιμαζόμαστε να βάλουμε στα χέρια του Ευρωπαίου πολίτη και αυτό με κάνει περήφανη. Αλλά θα πρέπει να είναι φιλικό προς το χρήστη, προσβάσιμο και αξιόπιστο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε σχετικά αυστηροί, να έγκυται στον τομέα των αρμοδιοτήτων, στο πατέρα των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις τεχνικές αυτές ε, απαιτήσει και νομίζω ότι πιο σημαντικό είναι ότι οι βουλευτές θα πρέπει να προετοιμαστούν να δράσουν από κοινού με τα άτομα που θα αναλάβουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Αυτό δεν υποσκάπτει τα δικά μας δικαιώματα. Μπορούμε από κοινού να το πετύχουμε με τους πολίτες. Θα πρέπει να κατευθύνουμε το μήνυμά τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε για να δημιουργήσουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή δημοκρατία. Ευχαριστώ κύριε Βουάλης. Άλλη αντιπρόεδρος. Τώρα έχει το λόγο η κύριε Ντιουράν. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο συνάδελφος κ. Χάφνερ μίλησε για κάποιες από τις προϋποθέσεις ούτως ώστε η πρωτοβουλία αυτή να είναι αξιόπιστη και νομότυπη. Να σας πω Δύο λόγια για την άποψη τη οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή που είναι ενδιαφέρουσα και μπορεί να μα φωτίσει στην απόφαση που θα λάβουμε και, να υπογρα... και που υπογραμμίσει το ότι η συμμετοχική δημοκρατία λειτουργεί όταν ο καθένα έχει το ρόλο του. Η αιρετή, εκπρόσωποι από την μια μεριά του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αλλά και οι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών και οι μη οργανωμένοι πολίτε, για του οποίου η πρωτοβουλία αυτή είναι μια ένα καινούριο στοιχείο. Υπογραμμίζω ωστόσο ότι το άρθρο 11 προβλέπει και την δυνατότητα διαρθρωμένου και οργανωμένου διάλογου με την κοινωνία των πολιτών. Τι προβλέπετε λοιπόν και αντιπρόεδρε σαν πρωτοβουλία όπως στον κοινωνικό διάλογο σχετικά. Θεωρείτε ότι ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί παράλληλα με αυτή τις πρωτοβουλίες των πολιτών. Σκέφτεστε δηλαδή να οργανώσετε έναν τέτοιο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών διαθρωμένο και διαθεσμικά. Για ένα λεπτό, ο κύριος Βαντάλεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χάρη στην πρωτοβουλία αυτή μπορούν να θέσουν τέτοιες πρωτοβουλίες οι πολίτες. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί απέχουν ακόμα πάρα πολλοί οι πολίτες από την Ευρώπη. Είναι μια καλή ευκαιρία για να μειωθεί η απόσταση με τους πολίτες. Να σας πω το εξή. Ο συνάδελφος Μάθεν Κάσλερ ξεκίνησε μια πρωτοβουλία στην οποία γίνεται έκκληση να τηρηθεί η Κυριακή ως ημέρα χωρίς εργασία, ημέρα μέρα της οικογένειας και της ε, ξεκούρασης. Θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε από κοινού όσο πιο πολλές υπογραφές γίνεται στην ε, Ολλανδία και θα ήθελα να σας καλέσω να υποστηρίξετε την πρωτοβουλία αυτή. Είναι σημαντικό αυτό και είναι σημαντικό να δείξει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και η Επιτροπή ότι είναι σημαντικά τα, είναι σημαντικές αυτές και προέρχονται από τον πολίτη και για τον πολίτη. Συνάδελφος Κολάσκα Μποβίνσκα, 1,5 λεπτό. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συνθήκη της Λισαβόνας αναβαθμίζει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τώρα έρχεται να συμπληρώσει αυτή την αναβάθμιση η πρωτοβουλία των πολιτών. Αλλά για να μπορεί να αποδώσει αυτή η ιδέα θα πρέπει να εκτελείται με κάποιες διαδικασίες με τις οποίες δεν υποβαθμίζεται και δεν υπονομεύεται το δημοκρατικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη φάση για την υλοποίηση πρωτοβουλία δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν έχει κάποια αρμοδιότητα. Στη κατά την προηγουμένη θητεία είχαμε ψηφίσει και εγκρίνει την πρόταση που θα ρύθμιζε την σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα τότε είχε πέσει το κοινό η πρόταση Κομισιόν, αλλά θα πρέπει και στην παρούσα φάση να περάσει η πρόταση αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί εμείς είμαστε οι εκπρόσωποι των ε, ψηφοφόρων, είμαστε το άμεσα εκλεγμένο όργανο, ενώ η Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο. Εάν επομένω η εκτελεστική, εξουσιοκριτικό όργανο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίψει μία πρωτοβουλία, τότε βεβαίω αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολύ άσχημες εντυπώσεις και οποιοδήποτε φορέα οποιοδήποτε με κυβερνητική οργάνωση η οποία βρίσκεται στην αφετηρία μιας της πρωτοβουλίας θα πρέπει να μπορέσει και να εξηγήσει και αιτιολογήσει και υποστηρίξει περί τίνος πρόκειται για κάθε πρωτοβουλία ακόμα και αν πρόκειται περί νομοθετικής πρότασης. Άρα θα πρέπει να εναρμονίσουμε τα εθνικά δίκαια σε σχέση με τις διαδικασίες που προβλέπουν τα, των πρωτοβουλίων. Γιατί αν υπάρχει πολυνομία τότε θα χαθεί η ουσία αυτή τη πρόταση. Για ένα λεπτό τώρα η κυρία Μπένοβα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών είναι ε, ένας θρίαμβος για τη δημοκρατία, διότι κατά αυτόν τον τρόπο εμπλέκεται ο Ευρωπαίος στις ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Επομένω, δεν μπορούμε να χαιρετήσουμε την πρότασή σα, αλλά τώρα θα ήθελα στη συνέχεια των είπε η κυρία Ζήτα Γκουρμάε, να, να, να, να τα επεκτείνω περισσότερο. Γιατί υπάρχουν πολλέ ερωτήσει, δεν έχουν λάβει απάντηση. Ένα από αυτά τα οποία σα ανέφερε είναι το τι θα γίνει με τι υπογραφέ. Πώ θα γίνεται η συλλογή των υπογραφών. Αυτό θα γίνεται από κάποιο κρατικό φορέα, θα γίνεται στο δρόμο. Μπά και καθ' τον τρόπο έχουμε φήμωση, περιστολή του, της ελευθερίας του λόγου. Επίσης, ε, από οικονομικής πλευράς, πώς θα καλύπτεται η πρωτοβουλία, θα είναι από τον κοινωτικό κορβανά, θα είναι από τον κρατικό κορβανά. Τι θα γίνεται ακριβώς, πώς θα, ποιος θα υποστηρίζει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας. Βεβαίως και έχει την, ε, το τίμημά της η δημοκρατία. Και επίσης θα πρέπει να δούμε το χρονικό πλαίσιο. Θα υπάρχει κάποια αποκλειστική προθεσμία μέχρι το τέλος της οποίας θα πρέπει να συλλεγούν οι υπογραφές. Επίσης θα πρέπει να δούμε προσοχή μήπως ανακατευτούν στη συλλογή υπογραφών κάποιοι που είναι κατά της Ένωσης. Ε, κυρία Χαρκίν, ευχαριστώ πρόεδρε. Δίσε τάχθην υπέρ ε, του ναι για τη συνθήκη της Λισαβόνας και διαφωνώ με τον συναδελφό μου. Ναι, υπάρχουν περιορισμοί, αλλά υπάρχει και δυναμικό και έχει σημασία να κάνουμε αυτό το βήμα για τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό. Έχω διευκολύνει και εγώ τις κινήσεις των πολιτών ε, ως προς τις διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης ε, ως προς τις ακροάσεις της Επιτροπής Αναφορών. Αλλά δεν αρκούν οι διαβουλεύσεις. Πρέπει να ακούμε τι λένε οι πολίτες ε, και να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις τους σε οποιοδήποτε νομοθετική πράξη εγκρίνουμε. Είναι σαφής προτεραιότητα των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Η πρωτοβουλία των πολιτών πρέπει να ισχύει από την αρχή μέχρι το τέλος. Πρέπει να είναι φιλική διαδικασία στους πολίτες ε, και να προωθήσουμε την ε, εικόνα της ε, να επικουρούμε τους πολίτες που επιθυμούν να αναλάβουν αυτή την πρωτοβουλία και να ξέρουμε πού μπορεί να δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πού όχι για να μην θα για δημοκρατικό έλλειμμα και να μην διωγγώνεται ο θυμός των πολιτών. Αν συλληφθούν οι υπογραφές παραδείγματος χάρη των πολιτών και κριθεί ότι ένα θέμα δεν είναι της αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα πρέπει να είμαστε προδραστικοί και ε, για να μην αποδυναμώσουμε την πρωτοβουλία, ας μην υποσχόμεθα περισσότερα από αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε. Ε, και πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή όταν αυτό το νέο μωρό, ας το θέσουμε έτσι, κάνει τα πρώτα του βήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αν λαμβάνω εγώ την Προεδρία της ε, Συνεδρίασης στα Ουγγρικά. Για ένα λεπτό λοιπόν η κυρία Λίχτενμπέρκερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι. Κατά τη διαμόρφωση αυτού του μέσου έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη γιατί οι ελπίδες των πολιτών που σκέφτονται ευρωπαϊκά νομίζω θέλουν και όσοι θέλουν να προχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα απευθύνονται σε μας. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη εκείνα που προδιαγράφονται. Δηλαδή να αποφύγουμε η πρωτοβουλία αυτή να μην γίνει ένα τείχος των δακρύων απλά χωρίς ε, να έχει αποτελέσματα. Οι ενεργοί πολίτες περιμένουν το αποτέλεσμα εάν είναι πολύ υψηλό το όριο θα απογοητευτούν πάρα πολλοί πολίτες. Σκεφτείτε, είναι πάρα πολύ μεγάλος κόπος να συγκεντρωθούν ένα εκατομμύριο υπογραφές για ένα θέμα. Εάν μετά δεν υπάρξει κάποια συνέχεια και χαθούν στο χαρτοβασίλειο, τότε νομίζω θα έχουμε βλάψει τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό τι θα κάνει η Κομισιόν εδώ πέρα. Αυτό για μένα είναι το βασικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για 1,5 λεπτό η κυρία Νεντέλτσεβα. Η πρωτοβουλία των πολιτών είναι ένας επιπλέον λίθος ε, για την ε, δημιουργία μιας πραγματικά δημοκρατικής ε, ευρωπαϊκής κοινωνίας και χάρη σε αυτήν μπορεί να ακουστεί περισσότερο η φωνή του Ευρωπαίου πολίτη όταν λαμβάνονται οι αποφάσεις και ελπίζω να ενισχυθεί και το αίσθημα που έχουν οι ναι. Ευρωπαίοι ότι ανήκουν σε μια ενότητα στην Ευρώπη γιατί έχει αποδυναμωθεί αυτή η αίσθηση. Έχει σχεδόν εκλείψει και πέρα από την πρακτική υλοποίηση της πρωτοβουλίας πρωτοβουλία μου φαίνεται ότι πρέπει να περάσουμε πάνω απ' όλα ένα πολιτικό μήνυμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ε, την βασική γραμμή αυτή τη πρωτοβουλία, δηλαδή να, γίνει, να πλησιάσει η Ευρώπη του πολίτε, ε, να προαγούμε την συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε συνέχεια κατά νου. Είτε μιλάμε για τον ελάχιστο αριθμό κρατών μελών από όπου θα προέρχονται οι υπογραφέ, η συλλογή των υπογραφών ε, ή ε, μιλάμε για το αν είναι παραδεκτές ή όχι οι αιτήσει. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να εμποδίζεται ο πολίτη από την κατάθεση μια τέτοια πρόταση. Να σα υπενθυμίσω ότι οι δαπάνε ε, τη επικύρωση μια υπογραφή από ε, συμβουλογράφο δεν είναι παντού ίδιες και τα καποια κάποια κράτη-μέλη που ε, δεν θέλουν να επιτρέψουν κάτι τέτοιο έχουν, επιβάλλουν υψηλό κόστο. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Να μην ξεχάσουμε επιπλέον ότι πρέπει να ενισχύσουμε το Κοινοβούλιο που είναι ο θεματοφύλακας τη δημοκρατική Βούλης των Πολιτών και εγγυάται την δημοκρατική διαφάνεια. Πρέπει να μετάσχει στη διαδικασία ε, της υλοποίησης αυτής της ε, πρωτοβουλίας. Γι' αυτό θα, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματική δημοκρατική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντερόσα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για μία από τις σημαντικότερες οικονομικές πρόοδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δύο τρίτα των Ιρλανδών υπεψήφισαν τη συνθήκη λόγω ακριβώς αυτού του χαρακτηριστικού. Για πρώτη φορά λοιπόν υπάρχει δυνατότητα μια τέτοια διεθνού πρωτοβουλία. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια όμω. Ποιο οργανώνει αυτέ τι πρωτοβουλίε και ποιο χρηματοδοτεί. Δεν πρέπει να το κάνουν οι επιχειρήσεις. Η Κομισιόν θα πρέπει να αποφασίσει αλλά Νομίζω πως εδώ πέρα θα, παίξει ένα, θα πρέπει να παίξει ένα σημαντικότερο ρόλο ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής για να κρίνει τι είναι παραδεκτό και τι όχι. Ο ελάχιστος αριθμός των κρατών που απαιτείται νομίζω θα πρέπει να είναι 7 και όχι 9 όπως προτείνει η Κομισιόν και πρέπει να επιμείνω πως το όριο του ενός εκατομμυρίου δεν θα πρέπει να ανέβει. και να γίνει ακόμη δυσκολότερο με το να έχουμε και ένα ακόμη ε, εμπόδιο με το να έχουμε μεγάλο αριθμό κρατών μελών. Επίσης θα πρέπει να μπορούν να γράφονται στο διαδίκτυο οι πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λούνατσεκ για ένα λεπτό η κυρία Λούνατσεκ. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την Ισπανική Προεδρία που ανέλαβε την ε, πρωτοβουλία να ξεκινήσει τη συζήτηση πριν από τα Τώρα συνεχίζω στα γερμανικά. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ την Κομισιόν που είχε αυτή την πρωτοβουλία και πράγματι ελπίζουμε μέχρι το καλοκαίρι να υπάρχει μια έτοιμη πρόταση. Σημαντικό είναι για τις προσδοκίες των πολιτών να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όπως και πάρα πολλοί συνάδελφοι βλέπω πως ανησυχούν όπως και εγώ ε, πως προσπαθούν οι νέες χώρες ε, να επιβάλλουν πάρα πολλά εμπόδια. Εγώ θα έλεγα να πάμε στις ε, πέντε χώρες και να μείνουμε δηλαδή στο 1 πέμπτο των χωρών και να είναι δυνατή η συλλογή και μέσω ίντερνετ. Επίσης η επίσημη εξέταση, η νομική εξέταση να γίνει στην αρχή και όχι όταν έχουν ξεκινήσει οι άνθρωποι να συγκεντρώνουν υπογραφές και θα πρέπει να υπάρξει στήριξη υπέχει μέσω μεταφράσεων. Αν συμβεί κάτι τέτοιο νομίζω θα τα καταφέρουμε να εμπλέξουμε τους πολίτες σε μια ισχυρή Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 1,5 λεπτό η κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω πως Ω προ την ε, υλοποίηση της συνθήκης Λισαβόνα, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι έχουμε στα χέρια μας ένα νέο αποτελεσματικό μέσο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και έτσι οι υπήκοοι των κρατών μελών θα μπορούν να ασκήσουν επιρροή στη δράση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης ε, και κατοχυρώνεται έτσι το δικαίωμά τους που συνιστά, όπως είπα, μέσω εκδημοκρατισμού αλλά βέβαια παρουσιάζει και κάποια μειονεκτήματα που οφείλουμε να εξετάσουμε. Πιστεύουμε ότι η προστασία των εθνικών συνταγμάτων ε, συνιστά προτεραιότητα. Πρέπει να κατοχυρωθεί αυτή η προστασία τους ε, και οφείλουμε να καταλήξουμε σε μία ισορροπία ε, και να μην χρησιμοποιηθεί το νέο μέσο ως πρόφαση που θα θέσει ένα αμφιβόλο την, το δημοκρατικό πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να διαλευκάνουμε λοιπόν ποιο ακριβώς θα είναι το πεδίο εφαρμογής πρωτοβουλίας ώστε να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες από πλευρά των πολιτών και των θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ για ένα λεπτό, Judith Μέρκης. Ναι, είμαι πολύ ικανοποιημένη με την πρωτοβουλία αυτή και αν δεν σας πειράζει τώρα θα μιλήσω Ολλανδικά για να εξηγήσω γιατί είμαι τόσο χαρούμενη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν θα λέει μόνο μία φορά στα πέντε χρόνια ποια είναι η απόψη του, αλλά μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζει ο πολίτης πότε μπορεί να έρθει εδώ πέρα να χτυπήσει την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε πρέπει να γίνει μια μεγάλη ενημερωτική εκστρατεία και βεβαίω εδώ πέρα το κρίσιμο είναι να ε, συνειδητοποιήσουμε πως ε, θα πρέπει να πάρουμε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σοβαρά το 1 εκατομμύριο υπογραφές. Και πράγματι όταν ένα εκατομμύριο όταν ένα εκατομμύριο πολίτες θέλουν να καταργηθεί το Στρασβούργο πρέπει να γίνει αυτό. Να τους ακούσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατόπιν. Κύριος Προβέρα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι αυτό το δικαίωμα πρωτοβουλίας που χορηγεί η συνθήκη στους Ευρωπαίους πολίτες θα οδηγήσει στο πλησίασμα μεταξύ των λαών και των λαών με την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ περισσότερο από, και θα αποδώσει πολύ περισσότερο από ό,τι απέδωσαν οι διάφορες ε, δάπανηρές ε, διαφημιστικές εκστρατείες. Αυτό θα προϋποθέτει και επιπλέον ενίσχυση της δημοκρατίας διότι οι πολίτες θα είναι αυτοί που θα προτείνουν άμεσα τους νόμους. Άμεση λοιπόν δημοκρατία η οποία συνοδεύει την κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτήν την ευκαιρία. Η Κομισιόν θα πρέπει να καταστήσει απλό και ευνόητο αυτό το δικαίωμα πρωτοβουλίας βοηθώντας τους πολίτες και συνοδεύοντάς τους από τη στιγμή της αρχής της διαδικασίας ορίζοντας σαφώς και τους όρους αποδοχής των προτάσεών τους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο Γιώργος Παπα-Νικολάου για ένα λεπτό Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συχνά αναφερόμαστε στην ανάγκη αύξησης της συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών, της ανάγκης να έχουμε πιο κοντά στους θεσμούς της Ένωσης, τους πολίτες όλων των κρατών μελών αυτό συζητήσαμε έντονα και στι τελευταίε ευρωεκλογέ, όταν σε πολλά κράτη-μέλη είδαμε ότι η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερω χαμηλή. Από τότε μέχρι και σήμερα μεσολάβησε ένα εξαιρετικό και σπουδαίο γεγονό που αλλάζει την ίδια τη δομή και τη λειτουργία τη Ένωση. Αναφέρομαι φυσικά στη συνθήκη τη Λισαβόνα, μια συνθήκη σημαντική, μια συνθήκη που κέντρο τη έχει τον πολίτη, που βασικό τη πυλώνα είναι πώ θα έρθουμε πιο κοντά στον πολίτη όλοι μα το κοινοβούλιο η επιτροπή το συμβούλιο και Εξειδίκευση αυτή τη αρχή είναι η πρωτοβουλία των πολιτών, το άρθρο 11, παράγραφος 4. Πρόκειται για μια σπουδαία ρύθμιση, για μια ρύθμιση η οποία είναι εξαιρετική, προάγει τη δημοκρατία, προάγει την πολιτική ισότητα, προάγει τη διαφάνεια. Το ζητούμενο βεβαίω είναι αυτή η ρύθμιση να εφαρμοστεί σωστά και να το δούμε στην πράξη και εδώ έρχονται οι προβληματισμοί εδώ πολύ σωστά τίθεται από όλους τους συναδέλφους η ανάγκη η διαδικασία αυτή να είναι αξιόπιστη να οριοθετηθεί ο ρόλος της επιτροπής ο ρόλος του κοινοβουλίου όλοι να μπορέσουμε να συλλειτουργήσουμε προκειμένου μια τέτοια σημαντική πρωτοβουλία των πολιτών αν συγκεντρωθούν μάλιστα υπογραφές να μην πάει στη συνέχεια χαμένη. καταλήγω λέγοντας το εξή, όλοι έχουμε ευθύνη να προβάλλουμε αυτή την πρωτοβουλία όλοι έχουμε ευθύνη να εξηγήσουμε το δικαίωμα αυτό που έχουν πλέον οι ευρωπαίοι συμπολίτε μα να του δώσουμε να καταλάβουν ότι μπορούν και οι ίδιοι να πυροδοτήσουν από την αρχή χωρί καμία άλλη μεσολάβηση διαδικασίε στο επίπεδο των θεσμικών οργάνων τη ένωση. και πάνω απ' όλα το μήνυμά μα αυτό να είναι καθαρό μέσα από μια διαδικασία απλή κατανοητή εύληπτη και αν μη τι άλλο λειτουργική για όλους λειτουργική για τους πολίτες λειτουργική για το κοινοβούλιο για του θεσμούς της ένωσης για τα κράτη μέλη για όλους τους φορείς που θα εμπλακούν στη διαδικασία. σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοέλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Προεδρεύω του, του Συμβουλίου, είπαμε πριν από λίγους ε, μήνες ε, ότι ποτέ δεν θα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Και τώρα όμως συζητάμε πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί και πώς θα εφαρμοστούν συγκεκριμένα κάποιες διατάξεις της. Και είναι πάρα πολύ σημαντική η συνθήκη της Λισαβόνας για την καταπολέμηση του δημοκρατικού ελλείμματος με την ενίσχυση του ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων και με, κυρίως μέσα από την πρωτοβουλία των πολιτών. Ελέγχεται έτσι η, τηρήση της αρχής της επικουρικότητας μέσα από αυτή την εξεκέλευτη πρωτοβουλία των πολιτών. Όπως είπαν και διάφοροι συνάδελφοι, κυρίως κυρίως ο κύριος Ντεβίγκο, θα ήθελα να επισημάνω ότι πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή ούτως ώστε να έχει ευρωπαϊκή διάσταση αυτό το μέσο για να εκφράζεται η πρωτοβουλία όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι κάποιων χωρών μόνο. Θα πρέπει να βρούμε επίσης μία λύση που να τονώνει την συμμετοχή, την καθημερινή συμμετοχή των πολιτών. Επίσης πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη σύνεση γιατί δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικοί υπερβολικά γενναιόδοροι. Αν βρούμε λύσεις που αποθαρρύνουν τελικά την συμμετοχή των πολιτών, θα προδώσουμε το πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας και την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Εμείς χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, την Ευρώπη των πολιτών, περισσότερη συμμετοχή των πολιτών ε, και μια δημοκρατική άσκηση του δικαιώματος και της ηθαγένειας των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ένα μισή λεπτό κύριο Σβέχ. Ευχαριστώ κύριε πίτροπε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που μπορώ να μιλήσω σήμερα για αυτήν την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία η οποία έρχεται να καλύψει το δημοκρατικό έλλειμμα ή τουλάχιστον θα προσπαθήσει να το καλύψει. Η δημοκρατία σήμερα βάσει των δημοσκοπήσεων βλέπουμε να περιορίζεται στα μάτια των πολιτών ως χώρος διαλόγου. Δημοκρατία όμως δεν είναι μόνο οι δημοκρατικές εκλογές. Δημοκρατία είναι η σχέση με τους πολίτες οι οποίοι είναι συνεχώς πιο παθητικοί, δεν συμμετέχουν στις εκλογές κλπ. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η συνθήκη της Λισαβόνας έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Και η προστιθέμενη αξία επίσης είναι αυτή η δυνατότητα πρωτοβουλίας των πολιτών. όπου μιλάμε για άμεση συμμετοχή των πολιτών. Πρόκειται για ένα σχέδιο Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Κάναμε ένα βήμα προς τα μπρος θα πρέπει να συνεχίσουμε στην οικοδόμηση αυτής της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και σε άλλους τομείς, για παράδειγμα στο διορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν ένα σωρό τομείς για τους οποίους τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να εκδημοκρατιστούν και να είναι και πιο δημοκρατικά. Ελπίζω αυτή η πρωτοβουλία να μας βοηθήσει να το κάνουμε. Ευχαριστώ κύριε Σβέρ. Ο κύριος Γιακολίνο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτροπή και συνάδελφοι, είναι μεγάλη ευκαιρία σήμερα να επικυρώνουμε εδώ μία νέα αξία, δηλαδή τη συμμετοχή του πολίτη η νέα δυνατότητα που δίνεται στον πολίτη για συμμετοχή με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Εγώ θεωρώ ότι λίγους μήνες μετά από τη θέση ισχύ της συνθήκης είναι πάρα πολύ θετικό να μιλάμε για αυτό το μέτρο. Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε με ακρίβεια τι εννοούμε ως σημαντικό αριθμό κρατών μελών. Θα πρέπει να έχουμε ένα κριτήριο το οποίο να συνδυάζει την παρόρμηση των πολιτών να συμμετέχουν και από την άλλη να δίνει το μέσο ε, για να καταστεί δημοκρατικό το μέσο. Χρειάζονται ελαφρές διαδικασίες, εύκαμπτες διαδικασίες. Εγώ αυτές τις τελευταίες εβδομάδες επισκέφθηκα πολλά σχολεία και είδα να υπάρχει μεγάλη διάθεση από τον κόσμο να ακούσει αλλά διαπίστωσα και τη συνέστηση που έχουν αυτά τα παιδιά ε, για την Ευρώπη το πώς αισθάνονται την Ευρώπη και πώς την ονειρεύονται θέλουν διαφάνεια, αντικειμενικότητα ούτως ώστε αυτό το μέτρο να είναι ένα μέτρο υπέρ της κοινωνίας. Γι' αυτό λοιπόν το Κοινοβούλιο ζητά να αποφασίσετε για ευέλικτες και απλουστευμένες διαδικασίες. Ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο. Ξεκινάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχω πάρα πολλά αιτήματα ομιλίας, δεν μπορώ να δώσω το λόγο σε όλους. Ο κύριος Μάρτιν Κάστερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ είμαι ένας από αυτούς που δημιούργησαν μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες πολιτών, δηλαδή για την προστασία της Κυριακής και μπορούμε τώρα να συζητήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να φέρουμε στην διαδικασία της πολιτικής εργασίας στην Ευρώπη για να έχουμε περισσότερη δημοκρατία κατά της κούρασης που επικρατεί γύρω από τα ευρωπαϊκά. Έχω όμως και δύο αιτήματα όταν θα πλησιάσουμε στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Πρώτα απ' όλα ως Ευρωπαίοι έχουμε τεχνολογία. Θέλω να σας παρακαλέσω το διαδίκτυο να γίνει το κατάλληλο μέσο έτσι ώστε με μια ηλεκτρονική υπογραφή η οποία ως γνωστόν είναι νομικά δεσμευτική να μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια πρωτοβουλία. Και δεύτερον εγώ θέλω να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Έχουμε τώρα δικαίωμα πρωτοβουλίας, αλλά στο μέλλον θα ήθελα να έχουμε και αποφάσεις των πολιτών, όπως την πατρίδα μου, την Βαβαρία. Υπάρχει και η δυνατότητα δημοψηφίσματος, εάν το ζητήσουν αρκετοί, και θα ήθελα να έχουμε στο μέλλον τη δυνατότητα αυτή στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Λίδια έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η δημόσια διαβούλευση για το θέμα αυτό τελείωσε και πόσοι έλαβαν μέρος 323 πολίτες πρέπει να ασχοληθούν επιτέλους ε, τα θεσμικά όργανα με αυτό το θέμα γιατί οι ελάχιστοι πολίτες γνωρίζουν ότι έχουν κάνει ένα τέτοιο μέσο στη διάθεσή τους. Μας δείχνει όμως πως τα πού πρέπει να πάει η Κομισιόν για την εφαρμογή της. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε σαφείς διατάξεις για τη συγκέντρωση των υπογραφών και το τι ισχύει στα κράτη-μέλη, π.χ. όσον αφορά την ηλικία. Μετά η εξάντε αξιολόγηση του παραδεκτού. Αυτοί που ξεκινούν μια πρωτοβουλία δεν μπορούν να νομίζουν πως ε, το παραδεχτό σημαίνει πως αυτομάτως η Κομισιόν θα κάνει και προτάσεις. Πρέπει να φροντίσουμε η πρωτοβουλία αυτή να οδηγήσει σε μια ευρεία συζήτηση για ευρωπαϊκά θέματα και αναμένω μια ανάλογη νομική βάση της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Κυρία Άντριου Μπράουνς κατόπιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η χρήση του δημοψηφίσματος ε, δεν είναι μια εξωτική εκδοχή της δημοκρατίας, είναι το πρωτότυπο. Να κυβερνούν οι πολίτες ε, και όχι να κυβερνούνται οι πολίτες. Ε, θα πρέπει ίσως να είμαστε και ευγνώμονες για την εισαγωγή του θεσμού. Αλλά δεν το νομίζω. Η Ευρώπη θέλει τη δημοκρατία όταν μπορεί να τη διαχειρίζεται και να έχει τα αποτελέσματα που επιθυμεί. Είχαμε τη δυνατότητα να συγκαλέσουμε δημοψήφισμα, αλλά μην ξεχνάτε τι έγινε με τα επιχειρήματα περί αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι σημαίνει αυτό? Περιορισμός της ελευθερίας ε, του λόγου και ακόμη και της σκέψης. Να πω και κάτι τελευταίο. Η δημοκρατία δεν σημαίνει κυβερνά ο λαός ε, με ένα συνεκτικό τρόπο, όχι να κυβερνούμεθα με αυθαίρετο τρόπο. Η μαζική μετανάστευση δυσχεραίνει τη διαδικασία και ολόκληρη η Ευρώπη τελικά δεν αποτελεί μια ενότητα, αντίθετα με αυτό που θα μπορούσε να είχε συμβεί. τέλο πάντων, ε, το μη χείρον βέλτιστο, αλλά πάντως είναι ε, κενό, κενή περιεχομένο αυτή η υπόσχεση περί πρωτοβουλίας των πολιτών. Ο σας ευχαριστώ. Η κυρία Έλενα Μπασέσκου τώρα για ένα λεπτό. Εγώ θεωρώ ότι η παρουσίαση αυτής της ε, πρωτοβουλία πολιτών της Ευρώπης είναι πάρα πολύ σημαντική και αποτελεί ένα βήμα πρόοδου για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Εγώ θέλω να σας πω ότι στη Ρουμανία από το 2004 μέχρι σήμερα είχαμε τρία δημοψηφίσματα και το τελευταίο αφορούσε στην ένωση των δύο βουλών και η συμμετοχή των πολιτών ήταν 51%. Συνεχίζω. Συγχαίρω λοιπόν εγώ την Κομισιόν για αυτήν την πρωτοβουλία, για αυτές τις ε, λαϊκές ετοιμιγορίες όπου θα οριστεί ο ελάχιστος αριθμός χωρών που θα πρέπει να συμμετέχουν όπως και ο ελάχιστος αριθμός υπογραφών. Πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσει να ισχύει αυτός ο κανονισμός, πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί όσο δυνατόν νωρίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σενάλοβα. Ευχαριστώ. Επίτροπε, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απολέσει την αξιοπιστία της. Αυτό φαίνεται από την χαμηλή συμμετοχή στις εκλογές, ε, διότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, κρίνουν ότι δεν μπορούν να επηρεάσουν τα πράγματα και γι' αυτό καλωσορίζουμε τη νέα πρωτοβουλία της συνθήκης της Λισαβόνας και επίσης την πράσινη βίβλο και τις διαβουλεύσεις ε, που γίνονται τώρα σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας. Συμφωνώ με την πλειοψηφία των προτάσεων που γίνονται, αλλά για να επικουρήσουμε τους πολίτες θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να γίνει αποδεκτή η πρωτοβουλία από του πολίτε. Ορισμένοι περιορισμοί είναι υπερβολικοί. Παραδείγματο χάρη, ελάχιστο αριθμό κρατών μελών από όπου θα προέρχονται οι υπογραφέ ε, των ε, πολιτών. Το 1 τρίτο των κρατών μελών. Αυτή είναι η πρόταση επιτάπητος, δηλαδή 9 κράτη-μέλη. Ε, είναι αποθαρρυντική αυτή η διάταξη και ουχή ρεαλιστική θα πρέπει να ε, πολεμήσουμε για το 20% του πληθυσμού της Ευρώπης ε, για να κάνουμε ένα σωστό βήμα, ώστε να εκπροσωπούνται σωστά οι περιφέρειες της Ευρώπης. Ο κύριος Σόγκορ. Ευχαριστώ. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικές δημόσιες συζητήσεις για ευρωπαϊκά θέματα, δηλαδή να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό κοινό. Η κοινωνία των πολιτών μπορεί να θέσει άρα εκείνα τα θέματα τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ευρωπαϊκά κόμματα. Τώρα, εγώ έχω να θέσω ένα ερώτημα. Είναι σημαντικό πριν ξεκινήσει η συλλογή των υπογραφών ε, να εκφράσει η Κομισιόν μία άποψη όταν ε, ξεκινάει η υπογραφή για το εάν ε, είναι παραδεκτή η πρωτοβουλία. Μην περιμένει οι άνθρωποι να μαζέψουν ένα εκατομμύριο υπογραφές και μετά τους πούμε δεν γίνεται γιατί θα απογοητευτούν με ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση πολίτε. Σα ευχαριστώ. Για ένα λεπτό. Η κυρία Μπλινκεβιτσούτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών και δίνει την δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες να ξεκινήσουν ε, με ένα εκατομμύριο υπογραφές μια τέτοια πρωτοβουλία. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο να συλλεχθούν τόσες υπογραφές όσον αφορά τώρα έναν αποτελεσματικό μηχανισμό αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και προσβασιμότητας οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τέτοιες προτάσεις με απλοποιημένη διαδικασία. Όμως με τη συνθήκη της Λισαβόνας ήδη ενισχύει, δεν εφαρμόστηκε ακόμα αυτή η διαδικασία, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα διασφαλιστεί η διαφάνεια για να μην πέσουν στα συμφέροντα και στην παγίδα των εταιριών οι πολίτες. Οπότε οπωσδήποτε αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού μέλλοντος και η Λιθουανία, η χώρα μου, θέλει ένα θεσμικό πλαίσιο. Οπότε ζητάω από την Κομισιόν να φροντίσει να τα εφαρμόσει αυτά το στομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά στο πλαίσιο του ΚΕΤΣΙΑΙ, για ένα λεπτό θα έπρεπε όλοι να αναγνωρίσουν ότι είναι πάρα πολύ θετική αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών ε, και στην Ιρλανδία μίλησαν για υφαρπαγή της εξουσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μια πραγματικά δημοκρατική απόπειρα αλλά ε, άλλο το να θεσπίζουμε κάτι και άλλο το να το υλοποιούμε. Υπάρχει, ελοχεύει ένας πραγματικός ε, κίνδυνος ε, κάποιες ομάδες συμφερόντων, τα λόμπι να καταχραστούν αυτή την πρωτοβουλία και γι' αυτό ο κύριο Εντερός έχει δίκιο ότι θα πρέπει να ε, αναβαθμίσουμε το ρόλο του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή. Βέβαια, υπάρχουν και πραγματικές ευκαιρίες ε, για τους ε, πολίτες και όπως είπε ο κύριος Κάστερ, θα έπρεπε να προωθήσουμε τις προσπάθειες που γίνονται και να αξιοποιήσουμε αυτή την πρωτοβουλία ούτως ώστε η 7η μέρα να είναι η μέρα του δημιουργού και όχι οποιαδήποτε άλλη μέρα. Σας ευχαριστώ και τώρα τελειώνουμε με τη διαδικασία του Catch the Eye και εξ ονόματος ε, του Συμβουλίου κ. Λόπες Γκαρίδο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ικανοποίηση για τη συζήτηση που έγινε και κατόπιν πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θέλησε να γίνει αυτή η συζήτηση για την πρωτοβουλία των πολιτών έγιναν πολλές τοποθετήσεις και διαπίστωσαν να υπάρχει απόλυτη ομοφωνία για την υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας η οποία αποτελεί προτεραιότητα για την Προεδρία του Συμβουλίου, την Ισπανική Προεδρία και θέλουμε να προχωρήσει γρήγορα. Με μεγάλη ικανοποίηση λοιπόν ακούσαμε και εμείς ε, την ε, εξαγγελία του κυρίου Σέρκοβιτς ότι θα παρουσιάσει στις 31 Μαρτίου τον κανονισμό. Ευχαριστώ την Κομισιόν για την ταχύτητα, για το ενδιαφέρον, για τον ενθουσιασμό με τον οποίο εξέτασε το θέμα και μπορούμε ήδη από τώρα να συνεχίσουμε, να, να ξεκινήσουμε όλη αυτή την νομοθετική διαδικασία την οποία σχεδόν όλοι όσοι μίλησαν θεώρησαν κατεπίγουσα και επιτακτική. Εγώ πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες υποστηρίζουν το μέτρο. Όλοι οι βουλευτές, ακόμη και όσοι δεν το υποστηρίζουν, πούμε, όπως ο κύριος Καμάλ, Λυπούμε που δεν είναι εδώ βέβαια. ο βουλευτής ο οποίος εξέφρασε τη φοβία ότι θα αποδυναμωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το μέτρο και να του πω ότι ίσα ίσα το αντίθετο θα γίνει, θα ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δύο βασικές ιδέες της Ένωσης θα ενισχυθούν, η δημοκρατία και το ανήκειν. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που θέλει να αντισταθμίσει αυτό το παράδοξο. Δηλαδή μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει όλο ένα και περισσότερες εξουσίες, μεγαλύτερη επιρροή, που επηρεάζει κάθε μέρα περισσότερο τη ζωή των πολιτών. Αλλά δεν έχει όμως ανταπόκριση όλο αυτό με την πολιτική συζήτηση που γίνεται στις χώρες μας. Και αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών που θα επεκτείνει το πεδίο των συζητήσεων για ευρωπαϊκά θέματα και όχι για τοπικιστικά θέματα διότι υποχρεώνει να έρχονται σε επαφή άτομα από διάφορες χώρες έχει πραγματικά ένα ευρωπαϊκό νόημα και είναι ένας τρόπος ενίσχυσης της δημοκρατίας αλλά και το αίσθημα του ανήκεινος πολίτη του ανήκειν δηλαδή στον Ευρωπαϊκό Δήμο που ανέφερε ο κύριος Κασίνη. Αυτό το ανήκειν ε, που ο κύριος Ραμόν Χαουρίγκη θεωρεί, ο κύριος Σόγορ θεωρεί πολύ σημαντικές και όπως είπε και ο κύριος Κέσλετ, αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να εφαρμοστεί. Διότι η ευρωπαϊκή πολιτική αγωγή αναπτύσσεται μόνο όταν εκτελείται, όταν μπαίνει στην πράξη. Και αυτό θα πρέπει να συμβεί από τη στιγμή που θα αρχίσει να ισχύει αυτό το μέτρο. Ευχαριστώ την Κομισιόν, ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θεωρώ ότι θα εξετάσει με ιδιαίτερη σοβαρότητα, με αυστηρότητα, αν και ο κύριος Γιακολίνο αναφέρθηκε στις γρήγορες ε, διαδικασίες για να μπορέσει δηλαδή να ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία το νωρίτερο δυνατό, και την κυρία Μπασέσκου η οποία είπε στην τοποθέτησή της ε, πόσο γρήγορα θα ήθελε να βλέπει να λειτουργεί το μέτρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υφυπουργέ. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Σεφτσοβίτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν καταπληκτική αυτή η σύνοψη της σημερινής ε, συζήτησης. Σας ευχαριστώ όλους ε, για την υποστήριξή σας και τις θετικές αυτές προσδοκίες σας ε, που συνδέονται με την πρωτοβουλία των πολιτών και με τα χαράς να σας υποβάλουμε την πρόταση το ταχύτερο δυνατόν μετά την έγκρισή της. Λόγω χρονικού περιορισμού σήμερα και λόγω του ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί η πρόταση δεν μπορέσαμε να υψέλθουμε σε λεπτομέρειες αλλά είμαι ευγνώμων που άκουσα τις απόψεις σας διότι απηχούν τη φύση και την ποιότητα των απόψεων που έχουμε συλλέξει από τους πολίτες προετοιμάζοντας αυτή την πρωτοβουλία. Για πάρα πολλά πράγματα συμφωνούμε. Ε, ένα από αυτά είναι η διαφάνεια. Σας διαβεβαιώ ότι ε, προσπαθούμε να βρούμε μια λύση που μέσα από την καταγραφή της πρωτοβουλίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κατοχυρώσει ε, την επιτυχία του επιτεύγματος. Να δούμε ακριβώς πώς θα χρηματοδοτηθεί για να διαπιστώσουμε αν πρόκειται για μια αυθεντική πρωτοβουλία των πολιτών, μια αυθεντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αν θα συγκεντρώνει δηλαδή όλα τα απαραίτητα στοιχεία ούτω ώστε να ε, στεφθεί με επιτυχία αυτό το νέο μέσο. Για την ε, πρακτική εφαρμογή συμφωνούμε όλοι. Θέλουμε να είναι φιλικό προς τους χρήστες ε, το νέο σύστημα. Δεν θέλουμε οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν την αίσθηση ότι θα ακολουθήσουν μια ιδιαίτερα επαχθή διαδικασία για να συλλέξουν, για να προσυπογράψουν μια πρόταση ε, θα διερευνήσουμε τις δυνατότητες και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής που χαρακτηρίζουν τον αιώνα μας. Είναι σαφές ε, ότι έχουμε διαφορετικά συστήματα εξακρίβωσης ε, της υπογραφής ανάλογα με το κράτος μέλος και μία από τις απαντήσεις που σαφώς προέκυψαν από τη διαβούλευση είναι ότι οι πολίτες επιθυμούν μία ομοιομορφία ως προς την εξακρίβωση και τη συλλογή των υπογραφών και ταυτόχρονα ε, τα κράτη-μέλη μας πέρασαν ένα σαφές μήνυμα ότι δεν πρέπει να είναι υπερβολικά βαρύ, υπερβολικά περίπλοκο το νέο σύστημα για τις εθνικές αρχές ε, γιατί τελικά τα κράτη-μέλη θα επιφορτιστούν με την εξακρίβωση ε, των ε, υπογραφών που θα συλλεχθούν για την πρωτοβουλία να εξακριβώσουν δηλαδή αν είναι γνήσιες οι υπογραφές των πολιτών. Άκουσα τις εκκλήσεις σας με προσοχή μου ζητήσατε σαφέστατες διαδικασίες μόλις ε, ε, μετά τη συλλογή των υπογραφών όταν κινηθεί δηλαδή η διαδικασία της ε, πρωτοβουλίας. Στην πρότασή μας θα υπάρχουν σαφή χρονοδιαγράμματα, σας διαβεβαιώ, σαφή χρονοδιαγράμματα βάσει των οποίων θα πρέπει να δράει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν στεφτεί με επιτυχία μια τέτοια πρωτοβουλία. Ακούγοντάς σας, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι το πλέον ε, περίπλοκο θέμα είναι αυτό του παραδεκτού των, ε, της ε, αίτησης των πολιτών πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες, να αντιμετωπίσουμε την αγανάκτηση των πολιτών, πώς να παραμείνουμε σοβαροί, να εφαρμοστεί με ουσιαστικό τρόπο αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις σε αυτά τα αντικρουόμενα αιτήματα, σε αυτά τα περίπλοκα ζητήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ταχθεί υπέρ της εναλλακτικής λύσης ε, που θα ε, υπερασπιστεί εξ αρχής τις ευρωπαϊκές αξίες. Ταυτόχρονα ε, θα θέλαμε να έχουμε μια σαφή εικόνα για την πρωτοβουλία των πολιτών για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ουσιαστικό δυναμικό για να τελεσφορήσουν οι προσπάθειές μας. Θέλουμε να αποφύγουμε τις καταχρήσεις ενδεχόμενες ε, καταχρήσεις αν έχουμε δηλαδή κάθε δύο εβδομάδες ε, τέτοιες ε, πρωτοβουλίες για ζητήματα που δεν αρμόζουν, που τελικά θα είναι θέμα μόνο του να εκδικαστεί αν είναι παραδεκτή η αίτηση ή όχι. Ε, δεν θέλουμε να ε, προαχθεί ε, το αρνητικό θεματολόγιο κάποιων ομάδων συμφερόντων και να υπάρξει κατάχρηση αυτής της πρωτοβουλίας. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τις ανάλογες απαντήσεις στο θέμα του παραδεκτού των ετοιμάτων των πολιτών. Τώρα για την κοινωνία των πολιτών έχετε δίκιο. Νομίζουμε ότι η καλύτερη απάντηση είναι αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών η ΕΟ και έχει διοργανώσει ε, έναν ε, πολύ ικανοποιητικό διάλογο για αυτό το θέμα και συζήτησα μαζί τους πριν από δύο εβδομάδες ε, και γίνονται δημόσιες διαβουλεύσεις μέσα από αυτές τις νομοθετικές προτάσεις που κάνουμε, ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιούμε όλο ένα και περισσότερο στο μέλλον ε, αδειμονώ να επανέλθω με την ε, συγκεκριμένη πρόταση για την πρωτοβουλία των πολιτών και ανυπομονώ να συνεχίσουμε το διάλογο τόσο ώστε αμελητή να εγκριθεί αυτό το τόσο ε, σημαντικό νέο νομοθετικό μέσο. ευχαριστώ πολύ. Εδώ πέρα λοιπόν τελειώνει η συζήτηση και αν επιτρέπετε περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήθειας διάταξης. Η κατάσταση στο Θιβέτ, δηλώσεις του Συμβουλίου και της